Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή μας, τους συνολότες, για τις επαφές που είχαμε για τον κύριο τοπκάι. Αποφασίσαμε χθες το βράδυ να ματαιώσουμε το ταξίδι μας στην Τουρκία. Για διάφορους λόγους. Ότι εκφράστηκε από την άλλη πλευρά ε, η διάθεση να μας υποδεχθούν μόνο εφόσον ήταν δεδομένο το αποτέλεσμα των των συνομιλιών. Δηλαδή προϋπόθεση ετέθη το άνοιγμα του κεφαλαίου 23. Μόνο αυτό. Επίσης μας είπαν ότι δεν μπορούν να συνομιλήσουν με ένα κοινοβούλιο το οποίο εγκρίνει ένα ψήφισμα και μπορεί το ψήφισμα ως προς το περιεχόμενο όταν είναι σωστό ή λάθος, αλλά είναι κυρίαρχο δικαίωμα ενός κοινοβουλίου να ε, συζητεί και να εγκρίνει οποιοδήποτε ψήφισμα θεωρεί σκόπιμο όταν είχαμε προγραμματίσει το ταξίδι αυτό, την αντιπροσωπή αυτό, αυτήν δεν υπήρχαν διαδηλώσεις και προβλήματα στην Τουρκία. Είχαμε τη διάθεση να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας, να συζητήσουμε τα διάφορα θέματα και να συζητήσουμε περαιτέρω την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εχθές, σε σχέση με την αντιπροσωπή αυτή, ανέλαβε μια συζήτηση με τον ε, ομόλογό του, του τουρκικού κοινοβουλίου και έτσι έγινε σαφές ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτή η αντιπροσωπή αυτή. Μια μικρότερη σύνθεση ομάδα απερίφθη ως πρόταση. Μια αποστολή από πλευρά ε, του Προέδρου του Κοινοβουλίου εκπροσώπων του επίσης απερίφθη. Προσπαθήσαμε λοιπόν σε κάθε επίπεδο. Είχα επαφές με τον Τούρκο Υπουργό των Ευρωπαϊκών Θεμάτων, οι οποίες επίσης δεν ήταν πολύ επικοδομητικές, χωρίς να θέλω να σας κουράσω με τις λεπτομέρειες, μπορώ να σας τα πω κατηδίαν, αλλά εάν ένας Γερμανός πρόεδρος κόμματος, μια Γερμανίδα καλύτερα πρόεδρος κόμματος βρίσκεται στο πάρκο Γκεζή και ε, εισπράττει δακρυγόνα, όπω η κυρία Κλάουδια Ροτ, και η απάντηση του Τούρκου Υπουργού των Ευρωπαϊκών Θεμάτων είναι «Ε, άμα φέρετε σαν τρομοκράτη, τότε θα έχει και την αντιμετώπιση που έχουν οι τρομοκράτε. Προφανώ αυτό εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ. Άλλα μέτρα επίση και αντίμετρα ε, απειλείται να επιβληθούν. Πρέπει να σα πω ότι είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Πιστεύω ότι η Τουρκία παραμένει πολύ σημαντικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις ε, περαιτέρω εξελίξεις εκεί και πρέπει να πούμε ότι όποιος σκοπεύει να γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει και να επιτρέπει τις διαδηλώσεις και να μην ρίχνει τους ε, διαδηλωτές στη φυλακή. Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει στη φυλακή δημοσιογράφους περισσότερους οποιοδήποτε άλλο κράτο και από ό,τι είχε δει τα τελευταία 75 χρόνια. Δεν το γνώριζα, το έμαθα όμως τώρα. Βλέπω ότι πρόκειται για πράγματα τα οποία πρέπει ρητά να καταγγείλουμε. Και αυτό βέβαια από την άλλη πλευρά δεν μπορεί και να σημαίνει ότι κόπτουμε, αποκόπτουμε τους δεσμούς. Αντιθέτως, θα πρέπει όποτε μπορέσουμε, όποτε μπορέσουμε να δούμε μια... Ε, βελτίωση της κατάστασης να αναλάβουμε και πάλι τις επαφές. Τώρα με ένα ματαιώνεται αυτή η αποστολή, αυτή η αντιπροσωπεία, αλλά ευκαιρία δοθήσεις θα επανασυνδεθούμε, θα επανασυνδέσουμε τις ε, επαφές μας και θα πρέπει να παρακολουθούμε και το θέμα της καταστολής των ε, διαδηλώσεων, της βίας, το χρονισμό αυτής της ε, καταστολής, αλλά βέβαια ε, με ό,τι χαρακτηριστικά η ε, περιγραφή και να δώσει κανείς δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η χαρακτηρισμή της τουρκικής κυβέρνησης για όλους τους διαδηλωτές συλλήφθηνων ότι πρόκειται περί τρομοκρατών. Έχουμε να κάνουμε με μια νέα γενιά, με νέους που διαδηλώνουν γιατί θέλουν μια κοινωνία φιλελεύθερη, γιατί θέλουν τα δικαιώματά τους γιατί θέλουν την προστασία του περιβάλλοντος και των πάρκων τους, γιατί θέλουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Πρόκειται για ένα ευρύτατο φάσμα ανθρώπων για τους οποίους, χωρίς βέβαια να μπορώ να πω ότι για όλους ισχύει αυτό, αλλά για τους οποίους σε πολλές περιπτώσεις τα, βλέπω ότι έχουν επιχειρήματα τα οποία δεν βρίσκουν σύμφωνο. Και νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την Τουρκία. Η πολιτική αυτή θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατό να προγραμματίσουμε περαιτέρω ταξίδια εν προκειμένου. Είχαμε ένα ταξίδι παλιότερα για την Ισλανδία το οποίο ματαιώθηκε, τώρα είχαμε για την ε, Τουρκία και πάλι χρειάστηκε να ματαιωθεί. Μήπως είναι τελικά επικίνδυνο να κανονίζουμε εμείς ταξίδια στους χώρες. Mm. Ας δω τώρα ποιος θέλει το λόγο, Sir Robert. Um, uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, βεβαίως. Ε, ε, επικροτώ την κρίση σας και τη θέση σας, αλλά κάτι με ανησυχεί, με προβληματίζει. Όπως είπατε στις παρατηρήσεις σας, είναι καλύτερα να κρατάει κανείς το διάλογο και την σύνδεση παρά να επιφέρει ρήξη διαιρωτώ με αν εσείς ε, και ίσως το θεωρήσατε αυτό μήπως να γράψετε στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας αναφέροντας ε, τις ε, ανησυχίες σας. Έχουμε μια διακεκριμένη επιτροπή με διακεκριμένο πρόεδρο και βεβαίως η επίσκεψη του Συμβουλίου είναι κάτι το σοβαρό. Το να γράψετε ίσως στον Πρωθυπουργό είναι αναγκαιότητα. Επίσης ανησυχώ προβληματίζουμε αν δεν θα, μήπως θα έπρεπε ε, να έχουμε μια ρήξη εφόσον παρουσιάσατε την περίπτωση όπως ε, το κάνατε σήμερα το πρωί Μήπως ε, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να σπάσουμε κάθε επικοινωνία. Είναι θέμα διαφοροποίησης χρειάς. Βεβαίως είναι να στην κρίση σας, δεν ξέρω. Διαρωτώ με αν όχι η πλήρης αντιπροσωπεία που θα πήγαινε ίσως μια μικρή ή εσείς ε, κάτι να κάνετε ακολουθώντας αυτόν τον προσανατολισμό ούτως ώστε ο Πρωθυπουργός να κατανοήσει ότι ε, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για μας όταν ένα μέλο μας τη χάνει αυτής της κακομεταχείρισης ε, και όταν υπάρχουν αυτές οι βιότητες είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό. Ε, θα πρέπει να θεωρήσει ο Πρωθυπουργό ότι αυτό είναι προσβλητικό για μας, αλλά θέλουμε να κρατήσουμε σχέση με την Τουρκία ε, προς όφελος του λαού και της χώρας και θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ε, η Ισλανδία και η Μουσκιώδης ε, εισηγητής τότε ε, και με την παρουσία του εισηγητή εξηγώ ότι πρέπει να πάμε εκεί. Ίσως μπορείτε να τους πείσετε, ίσως να υποβάλουν μια αίτηση. Ναι, ναι θα έλαβα ένα μέρο στην αποστολή στην, στην Ισλανδία, δεν πήγα από το 79 και έχω πολύ καλές αναμνήσεις από την επίσκεψή μου στην Ισλανδία, ίσως έπρεπε να ξαναπάμε. Αλλά θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ μαζί σας να γράψουμε μια τέτοια επιστολή στον Πρωθυπουργό ή στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, όχι σήμερα αλλά σε μερικές μέρες, να αφήσουμε ένα χρονικό διάστημα να περάσει και με μια εξήγηση Ίσως θα μπορούσαμε να δείξουμε ότι μας ενδιαφέρουν οι σχέσεις μας με την Τουρκία και το τουρκικό ε, κοινοβούλιο. Επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας θα μπορούσαμε από κοινού να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, αυτό που υπερέχει είναι ανησυχία σε δύο επίπεδα. Ανησυχούμε για την κατάσταση ε, στην ε, Τουρκία και η ανησυχία σε σχέση με τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι κάτι παραπάνω από εταίρος, είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αρχίσει με μια καλή είδηση διότι ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία των ε, πολιτών κινητοποιήθηκε γύρω από τον Γκέζι Πάρκ ε, με παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, πολύ καινούριε μορφές παρέμβασης ε, για την Ευρώπη ήταν μια κινητοποίηση των πολιτών που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αλλά αντιμετώπισε μια καταστολή πάρα πολύ σκληρή και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό ε, και σοβαρό είναι τα λόγια ενός ε, πρωθυπουργού ε, που έδειξε περιφρόνηση απέναντι στους διαδηλωτές που ήταν αλαζόν, που ήταν πάρα πολύ αυταρχικός, που ανέπτυξε την θεωρία της συνωμοσίας. Όλα αυτά μου φαίνονται ότι είναι, μας ανησυχούν και ρηπαίνουν τον πολιτικό διάλογο που θα μπορούμε να έχουμε με τις αρχές. Υπάρχει επίσης και η βία των αστυνομικών και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται ε, ακόμα και ε, η προσβολή και οι επιθέσεις στους ε, δικηγόρους, τους γιατρούς όσοι υποστήριξαν κατά κάποιο τρόπο τους διαδηλωτές και τους βοήθησαν και βοήθησαν το κίνημα αυτό του Γκέζι Πάρκ. Νομίζω ότι για όλα αυτά τα θέματα ήμασταν σαφείς στο ψήφισμά μας και όντως ε, η Τουρκία τόσο το κοινοβούλιο όσο και η κυβέρνηση θα πρέπει να μάθουν να ακούνε αυτού του είδους τις δηλώσεις. Δεν είναι κάτι το νέο εξάλλου, διότι στις εκθέσεις που υιοθετούμε κάθε χρόνο οι κριτικές εναντίον ε, της Τουρκίας για προσβολή, της και παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης, ελευθερίας του λόγου και του τύπου δεν είναι κάτι το καινούριο λοιπόν ε, και δεν είναι κάτι το καινούριο από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας ξαναδιαβάσουμε τις ετήσιες εκθέσεις και θα δούμε ότι είμαστε σε αυτά τα θέματα λεπτομερή ενδελεχής, σαφής και απαιτητική. Νομίζω ότι ο πολιτικός διάλογος, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να συνεχιστεί σε μια στιγμή κρίσης ακριβώς. Θα πρέπει να μπορέσουμε να πείσουμε για την σκοπιμότητα, για την χρησιμότητα των πολιτικών μας σχέσεων με την Τουρκία δείχνοντας πώς θα μπορούσαμε διαμέσου του διαλόγου να φανούμε χρήσιμοι, να φανούμε χρήσιμοι ούτως ώστε να καταλαγιάσει η κατάσταση και να υπάρξει μια διέξοδος από την κορυφή, από τα πάνω. Ε, μια προβλέπεται εξάλλου στις 27 και 28 Ιουνίου ε, μια συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και θα ήθελα να λάβει χώρα αυτή η συνεδρίαση για να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση αλλά θετική παραγωγική συζήτηση. Εδώ στις Βρυξέλλες θα έχουμε αυτή τη συνεδρίαση. Εγώ εξακολουθώ να σκέπτομαι αγαπητοί συνάδελφοι ότι θα ήμασταν πολύ πιο άνετοι, διότι θα ήμασταν πιο συνεπείς εάν εδώ και πάρα πολύ χρόνο δεν είχα, είχαμε δώσει στην Τουρκία και στις αρχές και κυρίως στον Υπουργό Δικαιοσύνη τον χάρτη πορείας για τα κεφάλαια 23-24 που θα μας επιτρέψουν να ασκήσουμε έναν μοχλό πίεση διότι διευκολύνουμε το παιχνίδι του Πρωθυπουργού που λένε «Α, είναι πολύ συμπαθητική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας ε, λένε τι πρέπει να κάνουμε», αλλά όταν πρόκειται να δράσουμε και να σταθμίσουμε τις ε, πολιτικές μας δεν κάνουν τίποτα εφόσον τα κεφάλαια παραμένουν κλειστά εγώ ε, θα ήμουν στο έργο μου πολύ πιο ήσυχη και άνετη και πιο συνεκτική και συνεπής αν ε, δεν μονομερός, ε, δεν κλείναμε το άνοιγμα των 23-24 και το κεφάλαιο 22 που είναι σημαντικό για την ειρηνευτική διαδικασία με τους Κούρδους. Μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι ένα θεμελιώδες διακύβευμα για την δημοκρατία την τουρκική την βάρινε πάρα πολύ το θέμα το κουρδικό και η διαδικασία συνεχίστηκε. Είδαμε ότι στην περιοχή των Κούρδων υπήρξαν πάρα πολύ λίγες διαδηλώσεις ε, δεν είναι λοιπόν οι άνθρωποι του ΠΚΚ που βρίσκονται στην πλατεία Ταξίμ, διότι οι περισσότεροι αντάρτες τώρα έφυγαν μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ειρήνης και θα πρέπει να σταθμίσουμε Ποιε θα μπορούσαν να είναι επιπτώσει πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι σημαντικό. Θα πρέπει εμεί με απαιτητικότητα και χωρί ταμπού να διαδηλώσουμε τις θέσεις μας και να είμαστε στεναροί στην βούλησή μας, να εμβαθύνουμε στο διάλογο αυτό και να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μας. Βεβαίως, οι διαδηλωτές δεν μας ζητούν να μπλοκάρουμε τα κεφάλαια 23 και 24. Ε, Θέλουν να είναι πολύ πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι διαδηλωτές. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνω τώρα τον κατάλληλο των μελετών. Πρώτον θα παρακαλέσω να είμαστε στο δυνατόν πιο σύντομοι στις παρεμβάσει μας για να μπορέσουμε και να κάνουμε ψηφοφορία με τον έχουμε αρκετό χρόνο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριος Πέτερλε, η Τουρκία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Τέτοιου είδους διαδηλώσει δεν είχε δει μέχρι τώρα ποτέ δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις διαδηλώσεις. Και ξέρετε, εγώ έχω δουλέψει στο παρελθόν σε θέματα χωροταξίας. Μπορώ να καταλάβω λοιπόν τι ζητούν οι ε, περιβαλλοντολόγοι, οι οικολόγοι αυτοί. Αλλά πάνω απ' όλα εδώ το ζήτημα και το διακύβευμα είναι το κράτος δικαίου. Εάν κατάλαβα καλά λοιπόν, έχει αποφασιστεί να μην αλλάξει η χρήση του πάρκου, του χώρου αυτού και να μην οικοδομηθεί. Ωστόσο, ακολούθησαν μετά την διθέτηση άλλου είδους διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, ε, προβληματισμοί. Και έτσι τώρα βρισκόμαστε ενώπιον πολλών διαδηλωτών διαφόρων ομάδων, μικρών ή μεγαλύτερων, από τους κομμουνιστές μέχρι τους ακροδεξίους. Ένα βρήκα το φάσμα διαδηλωτών. και βλέπουμε για πρώτη φορά να εκδηλώνεται η βούληση για έκφραση του πολίτη. Και για πρώτη φορά ζητείται υποστήριξη από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη έκφραση τη Βουλή των Πολιτών. Αυτό είναι μια νέα κατάσταση. Αρχικά, είχε ξεκινήσει ένα κίνημα από τη βάση, το οποίο ενδεχομένω να εξετάσει συνέχεια σε χειραγώγηση κάποιου βαθμού. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τον όρο τρομοκράτες για αυτές τις ομάδες των διαδηλωτών. Ας ε, σκεφτούμε λοιπόν πολύ προσεκτικά τι είδους διάλογο θα έχουμε από εδώ και μπρος με την Τουρκία και πώς μπορούμε να έχουμε τέτοιο διάλογο. Η αντιπαράθεση ασφαλώς είναι η χειρότερη λύση αν και υπάρχει ακόμη κίνδυνος να οξυνθούν τα πνεύματα και να προχωρήσει ακόμη περισσότερη αντιπαράθεση. Θα έλεγα λοιπόν να μην τίθενται όροι το να ορίζει, το να ορίζει προϋποθέσεις για το ταξίδι αυτό η τουρκική πλευρά δεν μου φαίνεται καθόλου επικοδομητικό. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση και ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τα κεφάλαια αυτά και βέβαια και η Μεκτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή να βοηθήσει ώστε να φτάσουμε σε μια καλή λύση. Ο Πρόεδρος, ναι, θα σας παρακαλέσω να είσαστε όσο δυνατόν πιο σύντομοι, 1,5 λεπτό θα σας περιορίσω. Κυρία Θεοχάρους, παρακαλώ. Αναρωτιέμαι, Πρόεδρε, αν πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από την Τουρκία γιατί αναγνωρίσαμε την γενοκτονία των Αρμενίων. Πρόεδρε, κάθε κίνηση προς την κυβέρνηση καλή θέληση από μέρου του Κοινοβουλίου που έχει επιδείξει πάρα πολλέ μέχρι τώρα θα ερμηνευτεί από του διαδηλωτέ ω πισόπλατο χτύπημα και οι διαδηλωτέ δεν διαδηλώνουν για το πάρκο αλλά για τι βασικέ και στοιχειώδει ελευθερίε του. Και εκείνο που ρηπαίνει τον πολιτικό διάλογο δεν είναι η συμπεριφορά η δική μα αλλά η συμπεριφορά των τουρκικών αρχών και η βαναυσότητα του απέναντι στον τουρκικό λαό. Έχω στα χέρια μου ένα γράμμα από τον πρόεδρο Σούλτ που ήρθε σήμερα και μα καλεί να συζητήσουμε για την προσβλητική συμπεριφορά του Μπαγής απέναντι στη συνάδελφο Ρενάτα Ζόμερ. Τώρα ακούω και για άλλη προσβλητική συμπεριφορά εναντίον ε, βουλευτήνα από τη Γερμανία. Έχω προσωπική πείρα από τη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου και άλλων πολιτικών και από τον τουρκικό τύπο. Πρόεδρε, εάν συνεχίσουμε να κάνουμε εκτόσεις, εκείνο που θα πετύχουμε στο τέλος είναι να απορροφηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από ένα στρατιωτικό μοντέλο. Γι' αυτό το λόγο η πρότασή σας για την υιοθέτηση του νορβηγικού μοντέλου είναι πέρα για πέρα αρκετή. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, νομίζω το είπαμε, το ξαναείπαμε, το είπατε και σήμερα, το είπαμε πάρα πολλές φορές ότι η Τουρκία για μας είναι σημαντικός εταίρος. Δική μου εκτίμηση πλέον είναι ότι αυτή η θέση περνά στην ιστορία. Θέλουμε ναι την Τουρκία να βρεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα ζήτημα. Ότι δεν πάει άλλο αυτή η συμπεριφορά της. Να προσβάλλει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσβάλλει ουσιαστικά καθημερινά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να κατευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς θα αποφασίσει, τι θα ψηφίσει, ποια θέση να πάρει. Προτείνω συγκεκριμένα. Σήμερα να καταδικάσουμε από αυτή την Επιτροπή, με τα όσα μας έχετε ενημερώσει, την πολιτική ευτογά... Να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μας στον τουρκικό λαό και στους διαδηλωτές και να δηλώσουμε ότι δεν είναι τρομοκράτες και βέβαια να στείλουμε πολιτικό μήνυμα ότι τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνει πλέον ανοιχτή και δεν πρόκειται να ανοίξει το κεφάλαιο 24 καθαρές κουβέντες για να προχωρήσουμε σοβαρά, υπεύθυνα και βέβαια να στείλουμε το μήνυμα που αρμόζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι στην κατηδία συνομιλία σας με τον κύριο Μπαγής ελέγχθηκαν πράγματα τα οποία, για τα οποία θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε κατηδίαν επειδή νομίζω δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα αυτή τη κατηδίαν ενημέρωση, αν έχετε εγκαλοσύνη, θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω δημόσια. Το δεύτερο που έχω να πω και αφορά τη συζήτηση που εξελίσσεται, εγώ θα συμφωνήσω ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία, στο αν δηλαδή στο τέλο εντάσσεται ή όχι, είναι πράγματι ασαφής. Ε, το μήνυμα που πάει προς την χώρα αυτή είναι ότι άλλες μεν χώρες το επιδιώκουν, άλλες κάνουν ότι το επιδιώκουν και άλλες κρύβονται πίσω από αυτές που πραγματικά το επιδιώκουν. Ε, αυτό είναι μια εικόνα η οποία ε, χωρίς καμιά αφιβολία δεν τους βοηθά. Όμως δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να συνδεθεί η στάση της τουρκικής αστυνομίας απέναντι στους διαδηλωτές με το αν έχει ανοίξει ή όχι το κεφάλαιο 23-24. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά τα δύο. Μπορεί να συζητηθεί το άνοιγμα των κεφαλαίων και να πάρει ο καθένας την τοποθέτησή του, αλλά δεν διασυνδέεται σε καμιά περίπτωση με, το, με την ε, σκληρή στάση της αστυνομίας απέναντι στο, στους διαδηλωτές. Ούτε υποθέτω εννοούσε κάποιος εδώ ότι αν, αν, αν ήταν ανοιχτά τα κεφάλαια η στάση της αστυνομίας θα ήταν διαφορετική. Το τελευταίο που, που θα ήθελα να πω είναι ότι ναι, οι, οι λύσεις έρχονται αν είναι κανείς καθαρός απέναντι στους συνομιλητές του. Και όσο καθαρή είναι η Τουρκία απέναντι σε εμά και μας τα λέει στα ίσα, όπως σας τα είπε εσάς ο κύριος, ε, ο, ο κύριος Μπαγής, ναι και το Κοινοβούλιο οφείλει να είναι πάρα πολύ καθαρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, καμιά φορά είναι καλό να μην εντείνουμε. Να μην οξύνουμε τα πράγματα μιλώντας ανοιχτά σε δημόσιες συνεδριάσεις. Πολύ ευχαρίστως να σας δώσω προσωπικός τις πληροφορίες που ζητάτε. Αλλά ας μην αφήσουμε περιθώριο για πιο μεγάλο θέαμα, ας πούμε, και, και φασαρία. Ξέρετε ότι εγώ ήμουνα υπέρ του ανοίγματο των κεφαλαίων. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο τώρα, αυτή την εβδομάδα, να γίνει αυτό το άνοιγμα. Και γι' αυτό προκύπτει με τις τελευταίες διαδηλώσει και την καταστολή ένα νέο, μια νέα εικόνα της Τουρκίας. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι υπέρ του να ανοίξουν τα κεφάλαια, αλλά χωρίς να ε, ξεχνάμε ποια είναι και τα δικά μας συμφέροντα και τι ζητούμε εμείς θα γίνει περαιτέρω προσπάθεια για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια Τουρκία που θα είναι πιο στενή δική μας σύμμαχος παρά κάποιον άλλον. Και αυτό εμένα θα με ησύχαζε πολύ περισσότερο από το να στρέψει το βλέμμα προς άλλη πλευρά η Τουρκία. Γιατί αυτό θεωρώ ότι υπαγορεύει και το δικό μας συμφέρον. Είτε είναι στο τέλος του δρόμου ως προοπτική η ένταξη ως πλήρους μέρους, είτε κάτι άλλο, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, η βασική μου θεώρηση είναι το συμφέρον, το μας είναι να είμαστε πιο στενοί συνομάχοι με την Τουρκία. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε και αργότερα. Τώρα κοιτάμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην ε, αντιμετώπιση της κρίσης. Τώρα πέραμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως που προβλέπει την ε, ε, ψηφοφορία στην έκθεση του κυρίου Μένεντες Δελβάλε. για την εταιρική σχέση με την Μαλαισία. Έχετε κάτι να πείτε κύριε συνάδελφε? Όχι. Τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Οι τροπολογίες 21 και 36 ψηφίζονται μαζί παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η τροπολογία 22 υπέρ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 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές. Οι σοσιαλιστές δεν βλέπω να συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Ή ε, τέλος πάντων πολύ υπογείως. 42 παρακαλώ υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Για την 42. Πέρα τις ψηφοφορίες. Απερίφθη. δεν βγήκατε αρκετά γρήγορα από το υπόγειο. «44 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 48 υπέρ, Τη 47 θέλετε να επελθεύσουμε. Πέρα τη ψηφοφορίες. 22 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. Θα ήταν πολύ κακό να είχα κάνει και πάλι λάθος. 48 λοιπόν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Θα παρακαλέσω τη σοσιαλιστική ομάδα, το κομμάτι εδώ προς τα μένα, να δραστηριοποιηθεί λίγο. Πέρα στις ψηφοφορίες. 20 υπέρ 24 κατά, απερίφθη ή 50. Στην 51 τώρα υπέρ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 Κύριος Κράισλ το είπε. Τα σχόλια δυστυχώς από την αίθουσα δεν ακούγονται. Ήδη το γμίγμα των συντακτών είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, ποιος λοιπόν υποστηρίζει αυτή την τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη Δέλτα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μια και ήταν τόσο πολλέ υπογραφέ, τόσο άλλο στο δεδομένο ότι θα εγκριθεί. Στη 16 παρακαλώ, υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται η υπαριθμόν 1 παρακαλώ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται η 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται πρώτη της Επιτροπής είναι τα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται είναι τα 2 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται τρία τη σύντα υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται. η Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της εκθέσεως. Πέρα της ψηφοφορίας. 44 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή μάλλον, εγκρίνεται. Äh, Και τώρα έχουμε την έκθεση από την αντιπροσωπή μας στη Γεωργία. Με επικεφαλής τον κύριο Λίμπορ Ρούτσεκ. Λίμπορ, αν θες να πάρεις το λόγο, παρακαλώ. So, colleagues, as you know, two weeks ago it was exactly... Συνάδελφοι, στις 7 Ιουνίου είχαμε μία αποστολή στην Γεωργία. Επτά μόν μετέβημεν και εκπροσωπούσαν πέντε πολιτικές ομάδες. Η αντιπροσωπεία λοιπόν δούλεψε μέσα σε μια καλή ατμόσφαιρα, σε καλό κλίμα. Συζητήσαμε με τις αρχές της Γεωργίας, συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και με τον Υπουργό των Εσωτερικών, τη Δικαιοσύνης τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, τον ε, Ombudsman και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να πούμε είναι πως η κατάσταση στη Γεωργία, όπως ανέφερα και χθε, ε, γνωρίζει μια μεταβατική περίοδο από ένα μονοκομματικό σύστημα σε ένα πολυκομματικό με τις φορές αυτή η μετάβαση είναι δύσκολη, η μετάβαση είναι περίπλοκη, η συνύπαρξη και η συμβίωση του Προέδρου με τον Πρωθυπουργό παραμένει σχετικά δύσκολη, υπάρχει πόλωση κοινωνική, το φθινόπωρο θα διεξαχθούν προεδρικές εκλογές Ένα από τα βασικά μηνύματα ε, που στείλαμε ήταν ε, να καταλαγιάσει η κατάσταση, να καθυσυχάσουν τα πνεύματα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τη Γεωργία για να περάσει αυτή τη μεταβατική περίοδο. Και τα όσα ακούσαμε αναφορικά με τον ευρωατλαντικό προσανατολισμό όλες οι όλα τα πολιτικά κόμματα, είτε βρίσκονται στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, τα μεγάλα πολιτικά κόμματα θέλουν να πετύχουν σε αυτό το έργο, δηλαδή την ευρωατλαντική ένταξη. Σε ό,τι αφορά τον διάσκεψη του Βίλνιους, θέλουν να πετύχει αυτή η διάσκεψη και να έχουν μια συμφωνία σύνδεσης αλλά και πρόθεση της συμφωνίας περί ελευθέρου εμπορίου. Μπορούμε να πούμε λοιπόν, συγκρίνοντας με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στους βασικούς προσανατολισμούς σε ζητήματα πολιτικής και διεξωτερικής. Ναι, υπάρχει αλλαγή σε ό,τι φορά τις σχέσεις και επαφές με την Ρωσία. Το συζητήσαμε με εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον Πρωθυπουργό Ιβάνη Τσφίλη και μας είπε πως η Γεωργία δεν έχει το σθένος ε, για να αλλάξει την κατάσταση. Μια νέα στρατηγική λοιπόν θα είναι να επικεντρωθεί στο να ανοικοδομήσουν την Γεωργία την ενίσχυση του πολιτικού συστήματος, ε, σε, του οικονομικού συστήματος, του κοινωνικού <clears throat> και αν ε, το κατορθώσουν να γίνουν ένα πρότυπο για την Απχαζία και για την Νότια Οσετία. Και αργότερα ενδεχομένως ο κύριος ε, Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αν υπάρχει κάποια αλλαγή με τη Ρωσία και εδώ βασίζεται στην ενίσχυση της κοινή των πολιτών και την έργο των ε, πνευματικών ανθρώπων στις μεγάλες πόλεις τότε ενδεχόμενα να θελήσουν να αλλάξουν κάποια πράγματα και να τα συζητήσουν αυτά τα ζητήματα. Προς το παρόν όμως δεν κρίνει ότι η Γεωργία έχει την ικανότητα και την ισχύ να αλλάξει το οτιδήποτε. Οι Γεωργιανοί επιθυμούν να συνεργαστούν με τη Ρωσία και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία το αποδεικνύουν π.χ. η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι ε, την υποκατάσταση ε, των εμπορικών σχέσεων. Ε, λοιπόν, η Ρωσία με όλα τα αυτά δεν τους κάνει πιο εύκολη τη ζωή στην κυβέρνηση του Ναντίον. Κρύβονται πίσω από διοικητικά θέματα από τον Υπουργό Εσωτερικών αλλά και από άλλες πηγές <clears throat> ακούσαμε ότι δημιουργούν, χτίζουν κάποια κάποια εμπόδια, κάποια τύχη σε κάποια χωριά. Βλέπουμε λοιπόν πως εδώ υπάρχει ανθρωπιστικό ζήτημα και από πίσω βρίσκεται το καθεστώς της Σετίας, της Απχαζίας κλπ. Αλλά αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν ως ανθρωπιστικής φύσης ζητήματα. Αυτοί οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκουν μπροστά τους το σύρματόπλεγμα δεν είναι τρομοκράτες, είναι πολίτες, είναι κάτοικοι των χωριών αυτών και κάτι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε την κατάσταση να αναφέρω κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις, διότι όπως σας είπα, ναι, υπάρχει μια μεταβατική περίοδος από το μονοκομματικό σύστημα στο πολιτικοματικό. Χθε συζητήσαμε την κατάσταση στις ε, τα διάφορα ιδρύματα Υπάρχει λοιπόν ευρεία συνένεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, διότι όταν έχουμε πολιτικοματικά συστήματα, οι καταστάσεις ξέρουμε ότι από εκλογές σε εκλογές αλλάζουν και αν η Γεωργία θέλει να προχωρήσει, θα πρέπει να πετύχει στις πολιτικές αλλά και στις άλλες μεταρρυθμίσεις. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Γεωργιανής Βουλής έθιξε διάφορα ζητήματα. Είπε ότι το 25% των εργασιών που διεξάγονται στο Κοινοβούλιο είναι ζητήματα τα επί των οποίων υπάρχει συνένεση. Συζητάνε η συγκυβέρνηση με την αντιπολίτευση και προσπαθούν να εξεύρουν λύσεις στα προβλήματα. τονίσαμε ότι αυτό απαιτείται όχι μόνο σε επίπεδο κοινοβουλίου, αλλά και σε επίπεδο προέδρου και πρωθυπουργού. Έτσι η κατάσταση δεν θα βγει εκτός ελέγχου. Το κοινό απαιτεί μια μεταρρύθμιση στο επίπεδο της δικαιοσύνης και δεν επιθυμεί να υπάρξει επιλεκτική δικαιοσύνη όπως ε, συμβαίνει τώρα. Αυτά είχα να πω. Ίσως ε, οι συνάδελφοι που ήταν παρόντες ε, στο ταξί αυτό να μπορέσουν να προσθέσουν κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Dziękuję bardzo. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Ρούτσε και Ήταν πολύ ε, ισορροπημένα παρουσιασμένη η έκθεσή του. Η αντιπροσωπεία μας είχε την ευκαιρία να συναντήσει όλες τις σημαντικές προσωπικότητες για την πολιτική ζωή της Γεωργίας. Θα πρέπει πάντως αυτή τη στιγμή να ε, τονίσουμε το ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και του Προέδρου της Γεωργίας πιστεύουν ότι δεν έχει μπει σε καλό δρόμο η χώρα, ότι έχει πάρει στραβό δρόμο και ως εκ τούτου. Όταν βλέπουμε να συλλαμβάνονται αντικαθεστωτικοί, Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είχαμε την ευκαιρία να συστήσουμε και με τον δήμαρχο της Τυφλίδας και, με τον και μάθαμε ότι ο πρόεδρος Σακασφίλη είχε πει ότι θα είναι ο επόμενος που θα μπει στη φυλακή. Άρα εκφράζονται αυτοί οι φόβοι ανοιχτά πλέον. Και άρα πρέπει δυστυχώς να ομολογήσω ότι η πολιτική κατάσταση είναι πολύ τεταμένη. Εχθές ανέφερα, επί παραδείγματι, ότι μόνο μία καλή ευκαιρία για συνομιλίες είχαμε, για επαφές σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και κανέναν άλλο διάβλο επικοινωνία. Πολλά είναι τα σχετικά μηνύματα. Επί παραδείγματι το γεγονό ότι ο Πρωθυπουργό και οι σημαντικότεροι υπουργοί δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και ότι η συνεργασία μεταξύ Πρωθυπουργού και Προέδρου είναι αδύνατη αυτή τη στιγμή. Η θητεία του Προέδρου σακασφιλη φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο σε μερικούς μήνες. Και η κατάσταση όπως έχει τώρα προφανώς δεν είναι καλή για την ε, Γεωργία και το μέλλον της. Δεν μπορέσαμε να συνομιλήσουμε τον Υπουργό των Οικονομικών επικεντρωθήκαμε μόνο σε θέματα συνταγματικής τάξης, νομικά ζητήματα. Και πρέπει να πούμε ότι στη Γερμανία, στην Γεωργία, συγγνώμη, ε, παρουσιάζεται και οικονομική ε, επιβράδυνση. Λόγω της ε, πολιτικής κατάστασης της χώρας παρουσιάζει σιγά σιγά επιβράδυνση η οικονομία μειώνεται η ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 50%, μειώνονται πολύ σημαντικά οι ξένες επενδύσεις τους τελευταίους μήνες, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση και περιπλοκή των ζητημάτων για τη Γεωργία. Ο κύριος Λάντσπερκης. Έχω μια παρατήρηση που δεν είναι μόνο ε, τυπική, αλλά περιλαμβάνει μερικές ενιολογικές ε, έννοιες ο συνάδελφος Ρούτσεκ ε, μίλησε για θέματα ε, διοικητικών συνόρων, σειρματοπλεγμάτων. Θα ήταν αντίθετο προς τη επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιείται η λέξη σύνορο. Δεν υπάρχουν σύνορα, είναι γεωργιανά εδάφη και είναι μια γραμμή κατάπαυσης του πυρός ε, που είναι εφικτή και κατανοητή. Ε, πώς εφαρμόστηκε, πώς θεσπίστηκε αυτή η γραμμή, το ξέρουμε πολύ καλά. Δεν είναι όπως ε, λέει η Ρωσία σύμφωνα με το δίκαιο της Νοτιού Οσετίας. Είναι ε, πάνω σε, ε, σε force majeure, σε ανωτέρα βία και δεν, και δεν τηρούνται τα πρότυπα κατά τη νομική έννοια. Ε, της, του διεθνούς δικαίου. Η ε, διοικητική ε, γραμμή μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν είναι σύνορο αυτή η διοικητική γραμμή. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνέδελφοι, ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας σας στην Γεωργία και θα ήθελα να πω μερικά λόγια και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ρούτσεκ για τον τρόπο με τον οποίο ε, ηγήθηκε της αντιπροσωπείας μας και για την αντικειμενικότητα της έκθεσης που μας παρουσίασε. Όπως πολλοί άλλοι στις εβδομάδες οδηγώντας στις εκλογές της κοινοβουλευτικές Έχω λάβει, κατακλείστηκα από εκθέσεις από όλες τις πλευρές που κατηγορούν οι μεν τους δε για ελιγμούς προσπαθώντας να επηρεάσουν ε, την εκλογική εκστρατεία και τις εκλογές και ήταν αδύνατο να καταλάβει κανείς ποιοι από αυτούς τους ισχυρισμούς είχαν βάση, ήταν αληθείς, αν ήταν υπερβολικοί ε, ε, ε, ισχυρισμοί αυτοί, λίγο υπερβολικοί, πολύ υπερβολικοί κλπ. Ήταν αυτό που μας εξέπληξε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων που είχαμε στην Τυφλίδα, οι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών, ε, το κόμμα του Προέδρου και τα άλλα κόμματα δηλαδή, παρουσιάστηκαν ως αθώα πρόβατα που δεν είχαν κάνει κανένα λάθος, δεν είχαν διαπράξει τίποτα το κακό, ως αν όλα να ήταν τελείως ειρηνικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, που δεν ήταν αυτή η περίπτωση και η αλήθεια. Είναι θαύμα που τα πράγματα δεν ε, εκτροχιάστηκαν, και η μετάβαση όπως γνωρίζουμε είναι κατά το μάλλον ή τον ειρηνική παρόλα που ορισμένη και εχθές εξέφρασα στην σύντομη παρέμβασή μου ε, και στις ερώτησεις στον επικεφαλής του Ρεπουμπλικού Κόμματος και πρόεδρο ε, του Κοινοβουλίου που είναι επικεφαλής της φιλελεύθερης ομάδας ότι ανησυχούμε, ανησυχούμε για την ε, σύλληψη του πρώην ε, Υπουργού Εξωτερικών που πριν από 8 χρόνια ήταν υπουργό Εσωτερικών. Είναι σημαντικό. Δεν ήταν υπουργός μια φορά, αλλά πριν από 8 χρόνια ήταν υπουργός Εσωτερικών. Ίσως είχε ε, ανάμειξη ε, στα αυτά που έκαναν ή δεν έκαναν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και νομίζω ότι είναι σημαντικό οι αρχές στην Γεωργία και το επισημάναμε αυτό, το επαναλάβαμε πολλές φορές στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον σημερινό Υπουργό Εσωτερικών, ε, στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ότι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα σενάριο του τύπου της Ουκρανίας εντός, εντός εισαγωγικών. Έχουμε προειδοποιήσει για το θέμα αυτό ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο σενάριο και ότι ότι ό,τι και να συμβεί δεν πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο σενάριο. Παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του σύνεγγης αλλά ταυτόχρονα δεν είμαστε αφελείς, τελείως αφελείς. Ε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Επιτρέψατε μου μερικές ε, παρατηρήσεις. Ε, ήμουν ε, μέλος της αποστολής αυτής, της διερευνητικής ο Λίμπορ ανέφερε ορισμένα πράγματα, αλλά αυτό που με εξέπληξε ήταν η συνάντησή μας με τα μέσα ενημέρωσης που δεν αναφέρθηκαν. Είχαμε ε, μια συνολική συζήτηση με τα μέσα ενημέρωσης, με τον Ombudsman, με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και αυτό που με εξέπληξε είναι ότι όλοι, όλα, όλες αυτές οι ομάδες, οι ανεξάρτητες και οι οργανώσεις όταν μιλούσαν για το παρελθόν μιλούσαν πάντοτε για την πολύ περιορισμένο χώρο για τις δραστηριότητες τους, πράγμα που σημαίνει ότι όταν ο Λίμπορ ανέφερε ότι υπάρχει μια, ένα μονοκομματικό σύστημα, μια κυβέρνηση μονοκομματική. Αυτό ε, περιόριζε πολύ τις δημοκρατικές δραστηριότητες των μέσων ενημέρωσης και των ΜΚΟ. Δεν θα αναφέρω εδώ όλες τις τεχνικές ε, λεπτομέρειες, αλλά δεν ήταν μόνον αυτό υπήρχαν πάρα, πολλές πολιτικές φυλακές στην πρώην κυβέρνηση και στο τοπικό επίπεδο, όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο υπήρχαν πολλές πολιτικά σημεία κράτησης. Περίπου 9.500 άτομα έχασαν την περιουσία τους, εκφοβίστηκαν από τις κυβερνητικές αρχές και πάρα πολλά άλλα πράγματα αναφέρθηκαν σε μια πολύ ανεξάρτητη συζήτηση την οποία είχαμε με αυτές τις οργανώσεις. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι δεν μπορώ να εμπιστευτώ τον πρώην πρόεδρο. Είμαι πολύ ειλικρινής ως προς το θέμα αυτό, διότι ο πρώην πρόεδρος θα έπρεπε να τα γνωρίζει όλα αυτά, τα όσα συνέβησαν, διότι ήτανε κάτω από την δική του ηγεσία που συνέβηκαν αυτόν. Ο, ο σημερινός πρόεδρος, ακόμη ε, σημερινός πρόεδρος μέχρι τον Οκτώβριο, με συγχωρείτε. Νομίζω ότι η νέα κυβέρνηση άνοιξε το χώρο, το δρόμο για την δημοκρατία, αλλά αυτό σημαίνει ότι ε, υπάρχει, υπάρχουν περισσότερες συγκρούσεις ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα σε αυτόν τον ανοιχτό χώρο και υπάρχουν τα πολιτικά κόμματα τα οποία είναι ανταγωνιστές που βρίσκονται ε, σε συνασπισμό, που βρίσκονται στην αντιπολίτευση και θα υπάρχει ένας αγώνας, μια σύγκρουση. Αυτό που προσπαθήσαμε εμείς να πούμε στη δική μας αντιπροσωπεία ήταν ότι η νέα κυβέρνηση, και αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα, εάν η πραγματική κυβέρνηση θα βρει το μέτρο, την σωστή ε, μεσαία γραμμή, το χρυσού κανόνα ε, και θα έχει την ικανότητα να αυτοπεριοριστεί σε ορισμένες δραστηριότητες αλλά αυτό δεν θα μπορεί να γίνει σε ολόκληρη την κλίμακα, διότι υπάρχει ένας πραγματικός πολιτικός αγώνας και θα πρέπει να δεχθούμε όταν έχουμε πραγματικές, πραγματικούς δημοκρατικούς θεσμούς να είναι αυτοί ανοιχτοί για τους αγώνες. Είναι αναγκαίο να υπάρχει βεβαίως ο αγώνας μέσα σε πλαίσιο μη βίας και σε πλαίσιο χρησιμοποίησης μόνο πολιτικών μέσων. Και αυτό είναι το θέμα. Και στην αντιπροσωπεία μας όλοι οι συμμετέχοντες ε, ευαισθητοποιηθήκαμε στο θέμα αυτό και κάναμε έκκληση στην κυβέρνηση να μην σταματήσει ορισμένες νόμιμες δραστηριότητες, αλλά όλες οι νόμιμες δραστηριότητες κατά της πρώην κυβέρνησης να είναι δίκαιες και αντικειμενικές. Και αυτό θα έπρεπε εμείς να προσέξουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν θα υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να πούμε ποιος είναι ένοχος ή ποιος δεν είναι ένοχος. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ περίπλοκη, αλλά αυτό που θα πρέπει ε, να παρακολουθήσουμε, να δούμε αν ε, οι δίκες θα είναι ε, δίκες και αντικειμενικές. Και νομίζω ότι ο νέος σύμβουλος του Πρωθυπουργού από την Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι θα κάνει τη δουλειά του με πολύ ικανοποιητικό τρόπο προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόβολ. Mam pytanie e, Κύριε Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση, ιδιαίτερα προς τον κύριο Ρούτσικ, αλλά και τον κύριο Λίσεκ. Και είναι η εξή. Ποιες προσωπικότητες της γεωργίας που παρουσιάζουν κοινωνικοποίηση, ε, δραστηριοποίηση, συγγνώμη, ε, όπως σε παραδείγματι οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο του διαμεσολαβητή. Αυτή είναι η πολύ σημαντική ερώτηση και η δεύτερη προς τον Πρόεδρο Μπρόκαλα και την Επιτροπή γενικότερα. Εμείς τι είδους ιδέες θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε προκειμένου να αποφύγουμε την κλιμάκωση της κατάστασης και των πιέσεων. Εάν δούμε ότι δεν αλλάζει η κατάσταση. Να αποφύγουμε την κλιμάκωση. Και εάν τώρα με νέα στοιχεία δούμε ότι ασκείται περαιτέρω πίεση προς την ε, αντιπολίτευση, προφανώς θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Τι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτή η επίσκεψη να μην είναι και η τελευταία μας, ώστε να αντιληφθεί η Γεωργία ότι πλησιάζει την κόκκινη γραμμή που έχουμε θέσει. Αυτό είναι το σχολείο μας. Όταν έχουμε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης στη φυλακή, πρέπει να μιλήσουμε και να μιλήσουμε με μία φωνή. Yes, ε, do you need the floor for Θέλετε το λόγο για να συναγάγετε συμπεράσματα. Μάλιστα. Ο κύριος Λαντσμπέργκης, ε, δεν ξέρω αν παρίσταται, μίλησε για τα διοικητικά σύνορα. Ποια είναι επίσημη έκφραση είναι ε, διοικητική συνολογική γραμμή. Και αυτό στην έκφραση χρησιμοποιούν όλοι στην Γεωργία, συμπεριλαμβανομένων και των Υπουργών. Στις συνεδριάσεις λοιπόν, στις ε, συνεντεύξεις τύπου, ναι, ε, τονίσαμε και είπαμε σαφώς πως εμείς στηρίζουμε την εδαφική ακαιρεότητα της γεωργίας, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν αυτά τα θέματα αναφορικά με την ε, διοικητική συνοριακή γραμμή. Πρέπει να βρούμε όμως κάποιο νόρο για να χρησιμοποιούμε και να προσδιορίζουμε αυτή την κατάσταση. Ο κ. Λατσμπέργκης μίλησε, έχετε να πω ότι Ακόμα και οι υπουργοί στην Γεωργία χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο της ε, διοικητικής ε, συνεργικής γραμμής. Μιλάνε για διοικητικά σύνορα. Ας φροντίσουμε λοιπόν ε, στον ελεύθερο χρόνο μας να βρούμε κάποιον όρο, κάποια έκφραση και να βοηθήσουμε τους γεωργιανούς φίλους εκτός μικροφώνου ο κύριος Λαντσμπέργκες, δεν τον ακούμε. Εν πάση περιπτώσει. Τα υπόλοιπα θέματα. Συνάδελφοι, δεν είναι μόνο η Γεωργία. Ουκρανία, Μολδαβία και άλλες χώρες στην Ανατολική εταιρική σχέση θα πρέπει εμείς ε, να δώσουμε ένα καλό θετικό παράδειγμα και να πούμε ότι στην δημοκρατία τα στρατηγικής φύσης ε, ζωτικά θέματα θα πρέπει να τύχουν συνένεση ε, σε όλο το πολιτικό τόξο. Ο κ. ρώτησε τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο Νομίζω πως ε, αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος μας ε, και να προσπαθήσουμε να καταλαγιάσουμε τα πράγματα διαδραματίζοντας ε, τον κατάλληλο ρόλο το όχι μόνο στη Γεωργία επαναλαμβάνω αλλά και σε άλλες χώρες. Ο κ. Φουρτάσεβιτς προ τριών εβδομάδων πήγαμε στη Μολδαβία ο ένας εκπρόσωπος του ΕΛΚ και ένας εκπρόσωπος της Σοσιαλδημοκρατικής Ομάδας μιλήσαμε με τους ε, ε, συναδέλφους μας εκεί και δύο μέρες αργότερα ανανέωσαν ε, την κυβέρνησή τους και την πολιτική ως εκ τούτου που ακολουθούσαν στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Πρέπει λοιπόν να διδραματίσουμε έναν θετικό ρόλο στο πλαίσιο της ε, ανατολική ε, γειτονία. Ίσως για κάποιους από τους συνέλφους μας ε, από το ΕΛΚ να είναι κάπως περίπλοκα τα πράγματα, διότι είχαμε συνηθίσει μια μόνο κομματική κυβέρνηση η οποία διοικούσε τα πάντα και ξαφνικά έχουμε μια νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Κόμματα τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν ανέλαβαν τη διακυβέρνηση. Αυτό νομίζω ότι είναι θετικό για την Γεωργία. Αλλά τώρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε από οποιοδήποτε κόμμα και αν προερχόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο να διαδραματίσουμε αυτόν τον ρόλο τον... Ε, του καταλαγιασμού και έτσι να επιτευχθεί η μετάβαση. Αναφέρθηκε ο κύριος Μιράβιτς. Χθες ε, ακούσαμε και από τον πρόεδρο της Βουλής ότι δεν είναι μόνο ο, δεν είναι μόνο ο αρχηγός της ε, αντιπολίτευσης, αλλά ήταν και υπουργό ε, εσωτερικών επί Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά από τις εκλογές δραπέτευσε από τη χώρα. Γιατί συνέβη αυτό, πρέπει να θέσουμε αυτό το ερώτημα. Χρειάζεται να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη χώρα. Όλα λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε να τα κατανοήσουμε και να μην κάνουμε σύγκριση Γεωργίας με Ουκρανίας, ε, την ε, σχέση του συμπεριφορά του Πρωθυπουργού με την στάση της κυρίας Τιμοσέγκο κλπ. Να επαναλάβω ότι η μετάβαση από μονοκομματικό σε πολιτικό σύστημα δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι απλό στις τελευταίες εκλογές υπήρξε η πιο ήρεμη ε, μεταβίβαση εξουσίας που έχει υπάρξει στην χώρα. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχουν ζητήσει το λόγο ο Σάιτ Βόλσκι και ο κύριος Τάνοκ. Δεν μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε τη συζήτηση. Αυτή είναι η πρακτική που ακολουθούμε τουλάχιστον διότι ο κύριος Μπουντούρ ε, περιμένει. Ξέρετε έξω έχει ωραία λιακάδα, λοιπόν ένα λεπτό έκαστος. Ένα λεπτό. Καμιά φορά υπάρχουν ε, σημαντικά θέματα ε, που απαιτούν να παρεκκλίνουμε από τους κανονισμούς. Είμαι ευγνώμων σε αυτά που ο Λίμπορ και άλλοι είπαν. Εάν βρίσκεται στην φυλακή ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, δεν υπάρχει δημοκρατική επιλογή. Με, με τον Γενικό Γραμματέα και με τους οικολόγους ΕΛΚ του ζήτησα να προσδιορίσουν μια κόκκινη γραμμή. Μια κόκκινη γραμμή είναι ανάμεσα στην δημοκρατία και στην μη δημοκρατία. Ο ηγέτης αντιπολίτευσης να είναι στη φυλακή, αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Όπως είπε ο κύριος Κόβαλ και άλλοι συνάδελφοι, έχετε δίκιο για τον Μαραμπισβίλη, αλλά οι φίλοι μας είναι στην κυβέρνηση, μπορώ να το πω αυτό. Ας ε, θεωρήσουμε να ζητήσουμε ε, κάθε ε, σύνδεση με μας αυτά τα κόμματα, διότι αυτό μας δένει τα χέρια αν δεν είναι αξιόπιτος ο Μυρασβίλη, ας ε, μην έχουμε αυτήν την σύνδεση, αυτήν την σχέση μαζί τους. Και η κόκκινη γραμμή θα πρέπει να είναι κοινή για ολόκληρο ε, το κοινοβούλιο μας, να μην υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι και να μην είναι ο αρχηγός της ε, αντιπολίτευσης. Ένα σχόλιο αυτό που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι όποιες σχέσεις και αν έχουμε με τον κόμμα στην κυβέρνηση, το κόμμα στην αντιπολίτευση, δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στο σύστημα δικαιοσύνης. Θέλουμε καλές σχέσεις με την Γεωργία και λυπούμε που βλέπω και μου φαίνεται ότι στη Γεωργία ε, η εισαγγελία, ε, οι ιδιοκτικές αρχές ε, και η δικαιοσύνη εξαρτάται από το ποιος βρίσκεται στην εξουσία. Αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο. Θα πρέπει οι ιδιοκτικές αρχές, οι εισαγγελικές, οι δικαστικές δεν είναι εξάρτητες από την κυβέρνηση και ξεπλάγινε χτες όταν ο, ότι είπε ότι ο, ο επικεφαλής του κοινοβουλίου, ο, πρόεδρος, ότι εκπροσωπεί την το, το κυβέρνηση. Όχι, δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Υπάρχουν μερικοί σαν αντιλήψεις περίεργες στην ε, Γεωργία. Όποιος είναι στο κοινοβούλιο προσπαθεί να ελέγξει το κοινοβούλιο, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, το δικαστικό θόμα. Θέλουμε ανεξάρτητο δικαστικό ε, σώμα. Αν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι στη φυλακή για οποιοδήποτε λόγο, δεν πρέπει να είναι στην φυλακή. Αν διώκεται για ποινικού λόγους, αυτό είναι διαφορετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, το επόμενο ε, θέμα θα το συζητήσουμε και κλεισμένων των ε, θυρών. Όσοι λοιπόν δεν είναι εξουδιωτημένοι να παραμείνουν στην αίθουσα παρακολούνται να αποχωρήσουν.